θα γίνει αύριο στις 10.30. Η επόμενη συνεδρίαση είναι αύριο 5η 19 Φεβρουαρίου στις 9 και επιτέλους μπορούμε να σβήσουμε